στην αρμόδια επιτροπή, δηλαδή στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Τέταρτη ανακοίνωση. Σας ανακοινώνω από την ομάδα ALDE και από την Γραμματεία των Μία έλαβα ε, κάποιες, ε, κάποια αιτήματα διορισμού στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ο, ο κατάλογος των ονομάτων αυτών θα δημοσιευτεί στα επόμενα πρακτικά και θα... Ε, ε, εγκριθεί ο διορισμός τους αν δεν διατυπωθούν ε, αντιρρήσεις πριν από το τέλος της σημερινής συνεδρίας. Τελευταία ανακοίνωση.